Συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Μερικοί από εσά μπορείτε να προτιμούσατε να ξεκινήσετε χωρίς τους σοσιαλιστές. <clears throat> Αλλά νομίζω ότι τώρα μπαίνουν οι σοσιαλιστές γιατί έρχονται από το διπλανό κτίριο. Μια στιγμή μονάχα λοιπόν, κάντε υπομονή και θα ξεκινήσουμε. Okay, I think we've waited long enough. Αρκετά τους περιμέναμε αυτούς τους σοσιαλιστές. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Εγώ είμαι προεδρεύων γιατί είμαι ίσως το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής αυτής στο Κοινοβούλιο. Όχι επειδή είμαι πιο μεγάλος από όλου να μην υπάρξουν παρεξήγησεις. Και είναι σύντομο το βασίλειό μου σε αυτή την ε, προεδρική έδρα. Απλώς πρέπει να εκλέξουμε πρόεδρο και αντιπροέδρους της ειδικής αυτής επιτροπής για την ε, χρηματοοικονομική κρίση βάσει του άρθρου 191 του κανονισμού. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος. Θέλω να θέσω το ερώτημα αν υπάρχει πρόταση για την Προεδρία της Επιτροπής. Μάλιστα. Υπάρχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον κύριο Βολφ Κλίντς θέλω να προτείνω για Πρόεδρο. Έχουμε άλλα ονόματα για τη θέση του Πρόεδρου. Όχι. Κύριε Κλίντς, συμφωνείτε με αυτή την πρόταση να αναλάβετε την Προεδρία. Ναι. Ναι, λέει ο κύριος Κλίντς. Εντάξει, μπορούμε λοιπόν διαβοής να εκλέξουμε τον κύριο Κλίντς. το χειροκροτήσατε πρωτού το πω κιόλα. μπορείτε να έρθετε να πάρετε τη θέση του Πρόεδρου. Liebe Kollegen, meine Αγαπητοί μου συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στην εκλογή των τεσσάρων, τέσσερων λέγω, αντιπρόεδρων. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριε Μπονσινιόρε, έχετε κάποια πρόταση για το, από την πλευρά του πολιτικού σας κόμματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την κυρία Ιβανόβα έχουμε να προτείνουμε. Apparently the, uh, it didn't work. Are you ready to uh, accept? Δέχεστε, αποδέχεστε την πρόταση αυτή εξ ονόματο της πολιτικής ομάδας. Άλλους υποψηφίους έχουμε. Έχετε κάνει δήλωση πόθεν όπως πρέπει. Έχετε. Ωραία. Η κυρία Ιβανόβα διαβοής επίσης προτείνω να εκλεγεί πρώτη αντιπρόεδρος. Συγχαρητήρια. Είστε η πρώτη μας αντιπρόεδρος. Ελάτε να καθίσετε δίπλα μου. We come now to, uh, Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο αντιπρόεδρο, Στίβεν Ιούς. Εσύ θα προτείνεις από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Α, την κυρία Λίζα Γιακονσάρη θα ήθελα να προτείνω. Πού κάθεται. Α, μάλιστα, η κυρία Λίζα Γιακονσάρη. Λάθος έκανε ο πρόεδρος. Αποδέχεστε το διορισμό σου. Κάνατε και εσείς την δήλωση υπόθεν έσχεση όπως πρέπει, μάλιστα. Ωραία. Is there any, is there any other candidate? Άλλον υποψήφιο έχουμε? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Και πάλι αβοήσει. So, congratulations, you are now the second vice. Συγχαρητήρια. Είστε η δεύτερη αντιπρόεδρος ελπίζω κατά τη διάρκεια των εργασιών να μάθω να λέω και το όνομά σας και να το προφέρω όπως πρέπει. Τρίτος αντιπρόεδρος, άνδρας ελπίζω αυτή τη φορά, από τους Πρασίνους. Σφεν. like colleague. Προτείνω τον συνάδελφό μου, Πασκάλ Κομφά, ο οποίος νομίζω θα συμβάλλει ιδιαίτερα στο έργο της Επιτροπής. Ε, ναι, κύριε Κανφέ. Είσαστε έτοιμος να δεχτείτε αυτό το διορισμό. Έχετε δηλώσει τα προσωπικά σας οικονομικά συμφέροντα κι εσείς. Α, τέλεια. Άλλοι υποψήφοι. Δεν βλέπω. Και πάλι σας προσκαλώ να εκλέξετε διαβοή στον κύριο Καμφέ. Ευχαριστώ. so Pascal Canfin is now the third chair. Ο Πασκάλ Καμφέ είναι ο τρίτος αντιπρόεδρος και ερχόμαστε στον τελευταίο, τέταρτο αντιπρόεδρο. Ο Νικόλαος Χούντις, ο οποίος θα παρουσιάσει τον υποψήφιο της ΓΚΟΕ. Τους ήδη εκλεγμένους αντιπροέδρους για την εκλογή σας, προτείνω τον Μιγγέλ Πόρτας για αντιπρόεδρο. Κάθε δίπλα σας κατά τύχη, μάλιστα. Είσαστε έτοιμος να δεχτείτε αυτή, αυτό το διορισμό. Έχω ήδη καταθέσει τη δήλωση οικονομικών συμφέροντων, λέει ο κύριο Πόρτα. Άλλοι υποψήφοι, όχι. Ε, φαντάζομαι ότι έχετε κάνει λοιπόν αυτή τη δήλωση, οπότε διαβοή καλό να εκλεγεί ω τέταρτο αντιπρόεδρο ο κύριο Πόρτα. So, you know, this is, this is a rather Ωραία, ήταν τυπικά όλα αυτά για να καθορίσουμε το Προεδρείο της ε, Επιτροπής μας. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω όλους που δεχθήκατε να προεδρεύω αυτή τη Επιτροπή. Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε με τη βοήθεια των τεσσάρων σοφών αντιπροέδρων καθώς και των συντονιστών, των σκιωδών συγητών, των ε, υπολείπων μελών της Επιτροπής μας να είναι επιτυχές στο έργο μας. Λοιπόν, η πρώτη συνάντηση των συντονιστών θα γίνει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο από τις 5.30 μέχρι τις 6.30. Θέλω λοιπόν να προσκαλέσω όλες τις πολιτικές ομάδες να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν τους συντονιστές τους ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. και όπου σε αυτή τη συνάντηση θα εξετάσουμε το σχέδιο εργασίας μας και τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Η πρώτη πλήρη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου 10 ως 12.30 το πρωί. Αυτά για σήμερα. <clears throat> και μου ζητήσαν επίσης να κάνω μια ανακοίνωση ότι σήμερα θα γίνει μια ανοιχτή συνάντηση των συντονιστών της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής με τον Τσάλι Μακρύβη που θα αρχίσει στις 11 στο άλλο κτίριο, στο ASP 3Ε2. Ε ε Όποιος θέλει να συναντήσει τον κύριο Μακρύβη λοιπόν και τους άλλους συντονιστές φυσικά μπορεί να πάει στο 3Ε2 στις 11 η ώρα. Ευχαριστώ και θα τα πούμε. Sorry. Sorry. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μου λέγουν ότι θέλει το λόγο Ρομπέρ Γκέμπελς. Θέλει το λόγο Ρομπέρ Γκέμπελς, παρακαλώ. Έχει κάθε δικαίωμα να μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρούμε ε, όλοι μας και εγώ προσωπικά και εσάς και τους αντιπροέδρους σας. Στην μερίσια διάταξη έχει και ένα πέντε που λέει τίποτα διάφορα εδώ. Και νομίζω ε, θα πρέπει σε αυτή την πρώτη συνεδρίασή μας της ειδική Έκτακτης Επιτροπής να σκεφτούμε λίγο πώς θα διαρθρώσουμε το πρόγραμμα εργασιών μας. Έχουμε μια καταπληκτική διοίκηση στο Κοινοβούλιο που πάντα προετοιμάζει τα πάντα και μας έχουν μοιράσει και έγγραφα, είχαν την πρόνοια, όπου ήδη έγραφε το όνομά σας ως πρόεδρος, πριν καν εκλεγείτε. Μάντης, μπράβο. Αλλά ε, έχουν καταρτήσει και ένα πρόγραμμα εργασίας για όλους τους επόμενους μήνες. Βέβαια, ε, ενδεικτικό το λέει η ρητά είναι αυτό, για να ε, βοηθήσει τους συντονιστές και να διευκολύνει τη δουλειά τους. Ελπίζω και να μην υπάρχει κανένας υπάλληλο που να γράφει ήδη την τελική έκθεση της ειδική μας Επιτροπής από τώρα. Και θα ήθελα να επιμείνω λοιπόν εξ ονόματος της ομάδας μου στην ανάγκη να γίνει ένας προβληματισμός σε βάθος για την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που θέλουμε να δώσουμε στις εργασίες της ειδικής του Επιτροπής. Εγώ έχω δεκαετή πείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμμετείχα και στις τέσσερις έκτακτες επιτροπές. Είχα μάλιστα την τιμή να προεδρεύω και σε μία. Και γνωρίζω πώς λειτουργεί το Ίδρυμα εδώ. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να κάνουμε μια θαυμάσια καταπληκτική έκθεση που θα πάει κατευθείαν στα σκουπίδια. Εκθέσεις για τη χρηματοοικονομική, πιστοτική και κοινωνική κρίση έχουμε τώρα δεκάδες επί δεκάδων στα κοινοβούλια. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα που να καταλήγουν στην νομοθετική μας εργασία, διότι είναι νομοθέτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή είναι η ισχύς μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο προσωπικά παίρνω το θάρρος να σας προτείνω να σκεφτούμε ίσως έτσι για αλλαγή να οργανώσουμε διαφορετικά τις εργασίες μας. η συγκήτριά μας βεβαίως είναι πάρα πολύ ικανή. Θα γίνουν και άλλες προτάσεις ε, από άλλους εξίσου ικανούς. Αλλά εάν θέλουμε πραγματικά οι προτάσεις μας να βγουν από ε, το κοινοβούλιο και προς τα έξω, μήπως θα έπρεπε να συνεργαστούμε με πανεπιστημιακούς υψηλού επίπεδου Θυμίζω σε όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα ότι στο Ευρωπαϊκό Κογκρέσο, στο Αμερικανικό των Ηνωμένων συγγνώμη, πριν από 10 χρόνια, είχε συστήσει ειδική επιτροπή γερουσίας και την αντιπροσώπου. Και ε, θέλησαν να ε, ε, συνεργαστούν με πανεπιστημιακούς υψηλού επίπεδου και βγήκε μια έκθεση λεγόμενη Μέλτσερ, η οποία είχε παγκόσμια απήχηση και ασχολήθηκαν όλοι οι μεγάλοι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με την έκθεση Μέλτσερ, ακριβώς διότι δεν περιορίστηκαν τότε στο να παρουσιάσουν μία έκθεση που έκανε απλώς οι πολιτικοί άνδρες. Εγώ είμαι πολιτικός και δεν απαξιώ καθόλου τους πολιτικούς, αλλά γνωρίζω ότι οι δικές μας προτάσεις κινδυνεύουν να ε, μπουν στο αρχείο εάν δεν ε, δώσουμε περισσότερο κύρος και περισσότερη ουσία. Εγώ μια πρόταση κάνω κύριε Πρόεδρε, δεν περιμένω να μου απαντήσετε τώρα, αλλά να το σκεφτείτε με τους ε, συντονιστέ σα και το Προεδρείο τη Δευτέρα για να ε, καταφύγουμε σε δυο τρει επαναλαμβάνω, αξιόλογους και υψηλού επίπεδου για να μας εμπνεύσουν οι πανεπιστημιακοί αυτοί. Μερσή ε. κύριε Γκέμπελς για τις παρατηρήσεις σας και τις συστάσεις σας. Σας διαβεβαιώ ότι πράγματι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πράγματι να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή στις εργασίες μας όλων αυτών οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν την εργασία μας και να μας δώσουν αποτελέσματα και συγκεκριμένες αναλύσεις. Επομένως δεν θέλουμε να έχουμε μια έκθεση η οποία δεν θα έχει καν αποτέλεσμα. Η δική μας Επιτροπή έχει συγκροτηθεί ως προσωρινή Επιτροπή, γιατί ήδη έχουμε στις μόνιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτροπές που ήδη έχουν εν μέρει αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και προφανώς πρέπει να έχουμε τους άριστους των αρίστων στην Επιτροπή μας για να μπορέσουμε να έχουμε τις χρωμοδοτήσεις τους και να έχουμε και διαγνώσεις αλλά και λύσεις για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο όπως είπατε και εσείς είναι ενδεικτικό. Μετά από τις συζητήσεις των συντονιστών μαζί με την εισηγήτρια, μαζί με τους γεώδεις εισηγητές θα μπορέσουμε να το εμβαθύνουμε περισσότερο το πρόγραμμα αυτό και να του δώσουμε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Παρακαλώ, έχει θέλετε το λόγο ο κύριος Μποργέζιο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Γκέμπελς, ήταν σοφά τα λόγια του, αλλά ήθελα να επιστήσω την προσοχή των μελών της Επιτροπής και της Προεδρίας κυρίως, του Προεδρίου μάλλον κυρίως της Επιτροπής, στην ανάγκη και όχι μόνο στη σκοπιμότητα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προσφορά συνεργασίας των ερευνητών, να μην ξεχάσουμε αυτούς τους λίγους μελετητές οι οποίοι, οι οποίοι είχαν προβλέψει την οικονομική κρίση. Τι και εγώ σας συμφωνώ με τα όσα ζήτησε ο Λουξεμβούργιος συνάδελφος και είμαι πεισμένος ότι χρειάζεται μεγάλη εξωτερική υποστήριξη πέρα από αυτήν των υπαλλήλων και των ικανοτήτων των συναδέλφων, γιατί γνωρίζω ορισμένους που πραγματικά είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι. Είναι μια κρίση εξαιρετικά δύσκολη που κατά την άποψή μου δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Έχουμε μια δημοσιονομική κρίση, χρηματοπιστωτική, έχουμε μια οικονομική κρίση. Ε, και φτάνει μια μεγάλη κρίση απασχόλησης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε στραμμένα τα μάτια ολόκληρου του κόσμου επάνω μας και κυρίως τα μάτια των χωρών της Ένωσης. Δεν μπορούμε να δίνουμε μόνο μια απάντηση ψηλού επίπεδου, ε, αφιψηλού. Ε, η δική μου ανησυχία είναι ότι πολλά πράγματα προσπαθούμε να τα κρύψουμε, να βάλουμε τα βρώμικα κάτω από το χαλί και να ξεμπερδεύουμε. Κατά την άποψή μου, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, πρέπει όλα αυτά να τα δούμε κατάματα και από την πλευρά του ΕΛΚ θα έχει η Επιτροπή αυτή όλη τη στήριξη που μπορεί να έχει για να αναλύσει καλύτερα και να μελετήσει καλύτερα και να δώσει όλες τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Όλοι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι και η φιλελεύθερη ομάδα θα σας υποστηρίξει πλήρως σε κάθε επίπεδο, σε κάθε βήμα. Συμφωνώ με τον κύριο Γκέμπελς, τον αγαπητό αυτό φίλο. Ρόμπερτ δεν πρέπει να υπερβάλλεις εαυτόν. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, έχουμε καταλήξει σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Αλλά αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπε στη... από τη μετάφραση, είπε ότι πολλέ από τι εκθέσει μα καταλήγουν στον καράθο των αχρήστων. Όχι. Ιδίω σε ό,τι αφορά την Οικονομική Επιτροπή τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κάνει καταπληκτική εργασία, έχουμε βρεθεί στην πρωτοπορία τη αντιμετώπιση πολύ δυσκόλων νομοθετημάτων και εξακολουθούμε να παίζουμε ένα σημαντικό. Ε, εντάξει, φταίνε οι διερμηνεί πάντα. <clears throat> Κλείνω λοιπόν, ε, κύριε Πρόεδρε, λέγοντα ότι ίσως πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα για να κάνουμε πιο λεπτομερή ανάλυση των ε, ε, επερχομένων ενεργειών και το τι θα κάνουμε στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Κυρία Ουλσκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Σουηδικά. Θέλω προφανώς καταρχήν να σας συγχαρώ για την εκλογή σας κύριε Πρόεδρε και εσάς και τους άλλους αντιπροέδρους. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος προηγουμένως. Γιατί έχουμε να αποθέσει πολλές ελπίδες σε αυτή την Επιτροπή. Θα πρέπει να εργαστούμε με ταχύτητα, θα πρέπει να εργαστούμε με υψηλή ποιότητα, να καταλήξουμε σε προτάσεις ποιότητος. Και ο λόγος ύπαρξής μας είναι πράγματι το γεγονός ότι οι μόνιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζονται η κάθε μία στο δικό της πεδίο του επιστητού. Ενώ η δική μας εντολή είναι διαφορετική και εμείς θα πρέπει να παίξουμε και τον ρόλο του συντονιστή κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των διαφόρων οπτικών γωνιών που έχουν να κάνουν με την κρίση. Όχι μόνο από την πτυχή της απασχόλησης, όχι μονάχα οι επιπτώσεις σε ό,τι αφορά στις μεθόδους παραγωγής. Σε ό,τι αφορά την αηφορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε την κρίση μονάχα υπό το πρίσμα των χρηματοοικονομικών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πτυχή την κοινωνική, την πτυχή της απασχόλησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα πιο αηφόρο υπόδειγμα στην κοινωνία μας. Θα πρέπει λοιπόν το πρόγραμμά μας να διατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να είμαστε αποκλειστικά και μόνο. Ένα εκτόπλασμα, κατά κάποιο τρόπο, μια προέκταση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξή. Κάνουμε τώρα πρώτη ανταλλαγή απόψεων σαν Επιτροπή. Ως Επιτροπή. Ακούω από αυτά που λέτε ε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαίρομαι γι' αυτό, το βρίσκω πολύ θετικό και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε όλη την ευκαιρία να κάνετε τις προτάσεις σας. Σήμερα όμως θα πρέπει να σας παρακαλέσω να περιορίσουμε σε ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό τις αποθετήσεις μας, διότι αλλιώς ξεπερνάμε το πλαίσιο που είχε προβλεφθεί το χρονικό. Έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Με χαρά να σας ε, το δώσω. Σφεν Γκίγορτ, Υπερβάνς Πασκάλ Κονφίν, ο κύριος Πόρτας, Κανάρ, Καμάρ, Βίκη Φόρτς και άλλη μια συνάδελφος μετά. Α, και ο κύριος Τόμας Μάν. Ναι, αλλά εδώ κλείνει ο κατάλογος για σήμερα των ομιλητών, διότι δεν θα προκάνουμε. Λοιπόν, επόμενος ο Σβέν Γκίγολτ. Πολύ σύντομα ο συνάδελφος από το Λουξεμβούργο έκανε μια πολύ επικοδομητική πρόταση. Είπε ότι πρέπει κανονικά να είναι προς το κοινό μας συμφέρον, να είναι όσο γίνεται υψηλή η προβολή του της, εδώ Επιτροπής. Είναι προφανές ότι θα βοηθήσει αυτό. Ε, δηλαδή να καλέσουμε κάποιους βασικούς εμπειρογνώμονες. Ε, βέβαια, ξέρω ότι είναι πολλά τα οικονομικά ζητήματα και η κρίση, αλλά καλό είναι να έχουμε τη συνεργασία κάποιων τέτοιων ε, εμπειρογνωμόνων. Είναι πολύ επικοδομητικό και δεν μπορούμε παρά να το υποστηρίξουμε. Merci. Ε, κύριε Μπερές, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Και θα έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε μαζί σας ε, στην Επιτροπή. Όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε ευκαιρία να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων στις προκαταρκτικές εργασίες μας ε, έχει προβλέψει τη σοφία της η διοίκηση στις 4 Νοεμβρίου να συνεδριάσουμε. Και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εντολή μας, ποια είναι η δυναμική της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν μπούμε στην ουσία των θεμάτων και των εργασιών. Ε, είχα και εγώ την ευκαιρία πάρα πολύ άτυπα να σας μιλήσω ήδη. Ε, θέλω να υποστηρίξω την πρόταση αυτή να έχουμε ένα είδος μόνιμη συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή, πέρα από τις προκηρύξεις που κάνουμε για μελέτες ε, ad hoc, θα πρέπει να έχουμε μια ομάδα πανεπιστημιακών, ε, εμπειρογνωμόνων, θα δούμε με ποια φόρμουλα θα γίνει και ποιο σχήμα, ε, για να μας υποστηρίζουν και στην ανάλυση μας πέρα από τις γνώσεις που έχει δική μας διοίκηση, για να μας βοηθήσουν στην τεκμηρίωση και την υποστήριξη. Είναι λίγο διαφορετική η πρακτική από αυτή που έχουμε ακολουθήσει στις τακτικές επιτροπές κοινοβουλευτικές και νομοθετικές του Κοινοβουλίου, αλλά είναι η η κατάσταση αυτή, έκτακτη προσωρινή επιτροπή με μία έκθεση που θα καλύψει όλη τη διάρκεια ζωής ε, της επιτροπής αυτής. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή, ένα επιστημονικό συμβούλιο να μας πλαισιώνει, να μας συνοδεύει και να απαρτίζεται ε, και να συσταθεί με τρόπο διαφανή. Ο καθένας να σέβεται τους κανόνες του Κοινοβουλίου βεβαίως. Το δίχως άλλο. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ευχαριστώ Περβάνς. Όπως πάντα κάνεις ε, πολύ χρήσιμες προτάσεις. Θα μπορέσουμε σίγουρα να συμφωνήσουμε γι' αυτό. Που είπες και εσύ και ο Ρομπέρ να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Νομίζω και όλοι Σμιτ λάθος κατάλαβε τελικά την πρόταση του Ρομπέρ Γκέμπελς. Ε, δύο σύντομε παρατηρήσει. Ο τρόπο με τον ε, οποίο ε, θα διοργανωθεί η εργασία να παράγει την διαχείριση ανά κομμάτια, ανά τμήματα, δηλαδή οικονομία, μετά οικονομικά και μετά κοινωνικά. Εδώ νομίζω πως πρέπει να κάνουμε το αντίστροφο. Ε, αν διατηρήσουμε ένα πρώτο πάνελ ε, για την ε, χρηματοπιστωτική κρίση, θα πρέπει το σύνολο, δεν θα πρέπει το σύνολο των παρεμβενόντων να είναι από τις τράπεζες, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα κτλ. Θα πρέπει και οι κοινωνιολόγοι και μακροοικονομικοί ε, να μπορέσουν να παρέμβουν, να παρέμβουν για τις ανισότητες, για να έχουμε πραγματικά μια οριζόντια εικόνα, πράγμα που θα μας αλλάξει από την εργασία που κάνουμε συνήθως σε νομοθετικές επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση στο προσωρινό έγγραφο εργασίας τελικά έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι θα ε, ξεκινούμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Να έχουμε όλοι την ίδια ενημέρωση, την ίδια γλώσση και αντίληψη. Αλλά η προσωρινή αυτή η έκτακτη επιτροπή ακριβώς γι' αυτό ιδρύθηκε, ε, συστήθηκε. Γιατί ξεπερνάει τα γνωστά πλαίσια και τα χρηματοοικονομικά και τα οικονομικά. Σήμερα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σημειώσουμε τις διάφορες ιδέες και θα το δούμε αυτό. Ο Βρετανός συνάδελφος. Αλλά προηγουμένως ο κύριος Πόρτας, το συγγνώμη. Ε, και εγώ πολύ σύντομα. Εγώ πιστεύω πως η πρόταση των σοσιαλιστών είναι ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να δούμε αν είναι εφικτή. Γιατί ταυτόχρονα πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο συνάδελφος ε, Κομφά. Να δώσουμε μια γραμμή εργασίας, δηλαδή μια ανάμεξη γνώσεων και ειδικοτήτων, που πιστεύω ότι επιβάλλεται. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σε αυτή την Επιτροπή είναι ότι στο πρόγραμμα των ακροάσεων θα πρέπει σίγουρα να εγγυηθούμε έναν μεγάλο, με μεγάλη διαφοροποίηση απόψεων για την ε, προέλευση και τη φύση της κρίσης που διανύουμε. Γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε δυσκολίες. Και ε, μια δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι και αφορά κάτι που θα ήθελα να σκεφτεί ο κύριος Πρόεδρος το περιβάλλον μας, το περιβάλλον αυτής εδώ της Επιτροπής, τοποθετείται περισσότερο στις ε, μεσοπρόθεσμες διαρθωτικές λύσεις. Όμως, μεταξύ, έχουμε και την Επιτροπή ΕΚΟΝ, που ασχολείται αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό πλάνο, με οδηγίες οι οποίες είναι απόλυτα διαρθωτικές για το μέλλον σε θέματα μελλοντικά. Άρα λοιπόν το βραχυπρόθεσμο και το μέσο πρόθεσμο θα πρέπει κάπως καλύτερα να τα κρίνουμε και πώς θα παίξουν όλα αυτά και πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να τα σκεφτούμε λίγο. Dear uh, uh, Σας ευχαριστώ. Μόλις ήρθε το μήνυμα ότι, έλαβα το μήνυμα ότι οι διερμηνείς έχουν προβλεφθεί μέχρι τώρα και πρέπει να φύγουν γιατί πάνε σε άλλη συνεδρίαση. Οπότε από εδώ και μπρος θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά.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 Okay.